Ε, καταρχήν θα συζητήσουμε την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον οξυοκομιακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις ενώσεις ΩΣΠΕΜ και ΕΠΣΟΥ. Η κυρία Λίν, η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν πέραν του ενός εκατομμυρίου ατυχημάτων που προκαλούνται από ο βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα τήσερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολύ ε, τραυματισμένοι πρέπει να περιμένουν για να γνωρίζουν εάν ε, υπάρχει ε, κάποιο πρόβλημα της υγείας τους ή κάποια μόλυνση η οποία να είναι πιο μακροπρόθεσμη ή όχι. Η, η υπόλοιπες επίσης ε, μολύνσεις είναι αρκετά σημαντικές. Ε, μπορεί να μολυνθούν ε, από την υπατήτηδα Β, υπατήτηδα Γ και από AIDS. Αν πάρετε την περίπτωση της Juliet Young που πέθανε το 2008 Επτά χρόνια αφού είχε μολυνθεί ε, από AIDS ε, την εποχή που έκανε μολυψία από έναν ασθενή σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου ε, προκλήθηκε όταν αυτή έκανε την εμολυψία. Ε, ε, ή ε, υπάρχουν ορισμένοι στις φυλακές οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία φυλακών όπου χρειάζεται να περιθάλψουν μολυσμένους φυλακισμένους ε, και ε, μία τέτοια νοσοκόμα ε, είχε συνάψει υπατήτητα Β. Εγώ είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό από το 2004 και είχα κάνει και μία έκθεση με τον Στίβεν Χιούς στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό. Το νοσοκομιακό και υγειονομικό προσωπικό ζητούν απεγνωσμένα τη βοήθειά μας και αυτοί οι οποίοι γνώρισαν τις νοσοκόμες αυτές και το άλλο υγειονομικό προσωπικό θα ε, συγκινήθηκαν προφανώς από τις εκκλήσεις τους και το 2006 ε, υπερψηφίσαμε ε, ένα ψήφισμα σχετικά με την προστασία του προσωπικού αυτού από τραυματισμούς που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα και ε, εκεί ε, βασίστηκε η ε, οδηγία 256 η οποία δεν υλοποιήθηκε τελικά ε, και γι' αυτό με το Steven Hughes ποτέ δεν απογοητευθήκαμε κάναμε πολλά ψηφίσματα φέραμε το θέμα στην Ολομέλεια επανειλημμένος και απαντήσαμε και υποβάλαμε ε, σε πάρα πολλές ε, ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο οπότε είχαμε φτάσει σχεδόν στο σημείο να επιτύχουμε αλλά η κοινωνική εταίροι τελικώς είχαν αποφασίσει να φτάσουν σε μία συμφωνία. Μία πλήρη συμφωνία πρέπει, έπρεπε να επιτευχθεί, πράγμα το οποίο έγινε το καλοκαίρι του 2009. Το ψήφισμά μου στηρίζει πλήρως αυτή, αυτή την συμφωνία και θα πρέπει το Συμβούλιο να αντιδράσει γρήγορα κατά τρόπον ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο χωρίς καθυστέρηση διότι ε, το υγειονομικό προσωπικό εξαρτάται από τις ενέργειές μας δεν μπορεί να κινδυνεύει συνέχεια και έχει φτάσει η στιγμή να δράσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χιούζ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα αυτό αφήνει το χρόνο στους εισηγητές να πάρουν τις θέσεις τους αντί να παραμένουν στην έδρα. Πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Καλό είναι να υπογραμμίσουμε το υπόβεθρο. Έξι χρόνια έχουν περάσει από τις πρώτες συναντήσεις ε, που κάναμε για το θέμα αυτό. Βλέπουμε και την αρμόδια επίτροπο εδώ σήμερα το πρωί. Δεν είναι όμως εδώ ο επίτροπος Σπίτλα. συχνά τον έχουμε επικρίνει, σήμερα όμως θα τον συγχαρούμε, θα τον είχαμε συγχαρεί αν ήταν, διότι προώθησε αυτή την ε, πρόταση για την πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα. Πολλοί τον συμβούλευσαν να μην δράσει. Πολλοί του έλεγαν ότι η οδηγία που εγκρίθηκε το 2000 για την προστασία των εργαζομένων από διάφορους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, μαζί με τα στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων της οδηγίας πλαίσιο του 99, αρκούσαν λοιπόν του έλεγαν όλα αυτά για την πρόληψη. Όμως, έχουμε ένα εκατομμύριο τραυματισμούς ετησίων και φάνηκε ότι βεβαίως κάτι πάει λάθος και χρειαζόμαστε ειδικά νομοθετήματα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό όπως ισχύει στη ΣΥΠΑ και ορισμένες αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας. Τελικά ο Επίτροπος συμφώνησε να δράσει και το 2008 διατυπώθηκαν κάποιες τροπολογίες στην υφιστάμενη οδηγία και <coughs> εστάλει αυτό το μήνυμα για την διατύπωση και Επίτευξη συμφωνία, η οποία είναι μεν καλή, είναι όμως και κάπως αμφίσιμη σε ορισμένα τη σημεία και γι' αυτό έχω υποβάλει μια τροπολογία την οποία έχει εγκρίνει και η Επιτροπή για την Απασχόληση, ώστε να έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές μαζί με την οδηγία για να διαβεβαιωθούμε για την ομοιόμορφη ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής στην εθνική νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Στηρίζουμε όλη αυτή την πρόταση. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ε, συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, η ρήτρα 6, που είναι και το πιο σημαντικό, η οποία έχει να κάνει με την εξάλληψη, την ε, πρόληψη και την προστασία, περιλαμβάνει κάποιες αμφισημίες, είναι κάποιες αμφίσιμοι ως προς ε, την αξιολόγηση επιπτώσεων και των κινδύνων μάλλον. Θα πρέπει να, να ξεκαθαρίσουμε αυτές τις αμφιβολίες που υπάρχουν στη διατύπωση της ρήτρα 6 και θα πρέπει η Επιτροπή να δώσει συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές τις οποίες θα πρέπει υποχρεωτικώς να λαμβάνουν υπόψη τους οι εργοδότες. Τραυματισμοί από βελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα είναι πολύ συνηθισμένοι. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται μία βελόνα σε έναν ασθενή, ελοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού και μόλυνσης, σοβαρής λίμωξης ή μόλυνσης ενός ε, εργαζόμενου στις φροντίδες υγείας και στην περίθαλψη γενικότερα. Ανεξάρτητα στοιχεία, στοιχεία ανεξάρτητων ερευνητών έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η χρήση ειδικών μηχανημάτων που ε, συμπεριλαμβάνουν είναι ήδη κατασκευασμένα με μηχανισμούς προστασίας θα ε, βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης. Είναι όλα αυτά απαραίτητα, αναγκαία. Και προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους μηχανήματα μόνο σε ορισμένες περιοχές ή μόνο σε ορισμένη κατηγορία ασθενών δεν ε, θα επαρκέσουν. Θα πρέπει να γίνεται ε, καθολική εφαρμογή αυτών των μηχανημάτων που έχουν ενσωματωμένου ε, μηχανισμού προστασία. Είναι πράγματα που γίνονται ήδη. Υπάρχει νομοθεσία ήδη στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και σε ορισμένε αυτόνομε κοινότητε τη Ισπανία και τι χρειαζόμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη ρήτρα 6, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια αμφισημία και θα πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε δημοσιεύοντας κατευθυντήριες γραμμές. Η προηγούμενη ομιλήτρια μίλησε και για τον ψυχικό τραυματισμό των εργαζομένων. Έξι χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα και έχω συναντήσει ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τη χρήση βελόνα σε ασθενή. Ένας γιατρός εγκατέλειψε την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος ε, κάποιος άλλος ε, έγινε οροθετικός επειδή μολύνθηκε μέσω της βολόνα που είχε χρησιμοποιήσει σε κάποιον ασθενή. Μολύνονται οι άνθρωποι, δεν το μαθαίνουν όμως αμέσως και ζουν επί μέσα σε αυτή την ε, δίνη, την ψυχολογική και την αβεβαιότητα. Πολλοί που συλλέγουν τα νοσοκομιακά απορρίμματα επίσης δεν μπορεί να μολυνθούν και δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία και δεν τυχαίνουν προστασία. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μειώσουμε, ελπίζω, ριζικά αυτό τον φοβερό αριθμό του ενός εκατομμυρίου τραυματισμών ετησίως. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον Επίτροπο Άντορ που έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Βούλιο για τις εργασίες του για το θέμα αυτό ιδιαίτερα την εισηγήτρια κυρία Λίν για την εξαίρετη προσπάθεια της για την γνωμοδότησή της για την πρόταση της Κομισιόν και για τις πολιετής προσπάθειές της για την βελτίωση της προστασίας του νοσοκομιακού προσωπικού. Ξέρω ότι είναι μακροχρόνια ανησυχία του Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα του 2005 του Κοινοβουλίου για την προώθηση της ασφάλειας των χώρο εργασίας κάλυσε για την αναθεώρηση της κοινοτική οδηγίας και ξανά τον Ιούλιο του 2006 υιοθετήσατε ένα ψήφισμα που καλούσε την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για τροποποιητική οδηγία της υφιστάμενης οδηγίας. Το Ευρωκοινοβούλιο μετά από αυτό το αίτημά του εξέτασε και τη νέα πρόταση της Κομισιόν σύμφωνα και με τις διεθνές προτάσεις της συνθήκης. Μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, δύο τομιακές ευρωπαϊκές οργανώσεις που δρούν στο νοσοκομιακό τομέα, η ΧΟΣΠΙΜ και η ΕΨΟΥ, διαπραγματεύθηκαν επιτυχώς μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ τους τον Ιούλιο του 2009. Όπως ξέρετε, η πρόταση του Κομισιόν έχει σκοπό να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τραυματισμοί από αιχμηρά αντικείμενα είναι από τα τις μεγαλύτερες απειλές στο νοσοκομιακό προσωπικό, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς όπως είναι τα επίγοντα περιστατικά ή τα χειρουργεία. Χαίρομαι γιατί το ψήφισμα σας αναγνωρίζει ότι η πρόταση της Κομισιόν ενσωματώνει τα χειρουργια χαιρομαι γιατι το ψηφισμα σας αναγνωριζει οτι σημεία του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου του 2006. Η Κομισιόν ή επιθυμούσε να συμπεριληφθούν στη συμφωνία τα σημεία αυτή. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι η θέση σε ισχύ αυτής της συμφωνίας θα είναι μια σημαντική συνεισφορά για την προστασία του προσωπικού στον υγειονομικό τομέα. Με τη συμφωνία αυτή και ελπίζουμε και την μελλοντική υιοθέτηση από το Συμβούλιο της προτινόμενης οδηγία, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομιακό και υγειονομικό τομέα θα τύχουν ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα έχουν πολιτικές, αξιολόγηση κινδύνου, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση και ούτω καθεξής. Τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία είναι ελάχιστες απαιτήσει, όχι μόνο είναι καλοδεχούμενα αλλά και απολύτως απαραίτητα. Πρόεδρε, κυρία Ισηγήτρια, μέλη, κλείνω ευχαριστώντας γιατί υποστηρίξατε την πρόταση της Κομισιόν και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα την υιοθετήσει λίγαν συντόμως. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Μπάλτασάρε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε, τα, οι τραυματισμοί από τα αιχμηρά αντικείμενα είναι από τους κοινούς κινδύνους που αντιμετωπίζει το νοσοκομιακό προσωπικό στην Ευρώπη και είναι μεγάλο πρόβλημα και για την κοινωνία και για την υγεία. Η παρούσα πρόταση της Κομισιόν έχει σκοπό να δώσει στο Συμβούλιο να ε, επικυρώσει την διμερή συμφωνία των δύο τομεακών οργανώσεων της Ευρώπης, την ΟΣΠΙΜ και την ΕΦΣΟΥ. Η συμφωνία έχει στόχο να δώσει μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους από τους κινδύνους τραυματισμών που προκαλούνται από εχμηρά αντικείμενα και χρησιμοποιούνται στον υγειονομικό τομέα. Είναι σημαντικό βήμα προόδου για την βελτίωση της ασφάλειας στο νοσοκομιακό τομέα και όπως όλοι ξέρουμε οι συνέπειες αυτών των τραυματισμών μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και να οδηγήσουν σε διάδοση ασθενειών όπως η υπατήτηδα ή το AIDS. Πρέπει να έχουμε μία ρεαλιστική και φιλόδοξη προσέγγιση στο πρόβλημα αυτό. Και θεωρώ σκόπιμο τα, γραφειοκρατικά βάρη, τα να μην είναι υπερβολικά εξαιτία αυτής της συμφωνία και να μην είναι ει βάρο της ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δρούν στο νοσοκομιακό τομέα, οι οποίες αλλιώς θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες για να σεβαστούν τους όρους της συμφωνίας. Επίση, υπάρχει η δυνατότητα, όπω προβλέπετε, για τα κράτη-μέλη, και να υιοθετήσουν διατάξεις, μέτρα και μέτρα πιο αποτελεσματικά από αυτά που περιλαμβάνονται στη συμφωνία για να προστατεύσουν τους εργαζομένους τους. Τέλος, ζητείτε από την Κομισιόν να προσέξει την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας και να μας ε, να ενημερώνει τακτικά το Ευρωκοινοβούλιο για την πρόοδο της εφαρμογής. Να έχουμε έτσι μια σωστή παρακολούθηση της συμφωνίας και να αξιολογήσουμε την πιθανή ανάγκη λήψης μελλοντικών μέτρων. Κύριος Τσέρκας, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να, να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Λίν για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην Επιτροπή μας, διότι μπόρεσε να συμφιλιώσει όλες τις απόψεις και να δουλέψει τόσο επικοδομητικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας συγχαίρω, Επίτροπε Άντορ. Είστε δεύτερη μέρα στα καθήκοντά σας. Έχετε ξεκινήσει πραγματικά με το δεξί. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά ήδη. Και προχωρείτε, βλέπω, και άλλη οδηγία και μια άλλη οδηγία το, για την χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η οδηγία αυτή έχει απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζουμε λοιπόν να λύσετε γρήγορα αυτά τα δύο προβλήματα τα οποία θα δώσουν ελπίδες ε, σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ και τη δουλειά του Επιτρόπου Σπίτλα για τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα, αυτό το νομικό μέσο αφορά πάρα πολλούς εργαζομένους στον τομέα της υγείας και είναι πολύ σημαντικό το εργαλείο αυτό για αυτούς τους ανθρώπους ε, θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα όλες αυτές τις λοιμώξεις και τις μολύνσεις από διαφόρους ιούς τους ιούς της υπατήτηδας ή του HIV και το καθεξής. Θα ωφελήσει λοιπόν όλους τους εργαζόμενους, αλλά θα ωφελήσει και τις οικογένειές τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, καλώντας συνεχώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να το ακολουθήσει και θα πρέπει να επενθυμίσουμε και τη δουλειά του κυρίου Χίουξ. Επιτρέψτε μου όμως να προβώ σε μια αξιολόγηση των λόγων για τους οποίους χαιρόμαστε σήμερα εμείς όλοι οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές. Καταρχάς, έχει τεράστια σημασία βεβαίως το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο ε, υγιούς χώρου εργασίας είναι ζωτική σημασία για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στις ε, πολύ θετικέ επιπτώσεις που θα έχουν τέτοιου είδους νομοθετήματα ε, για τους ε, εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Όμως, εξίσου ωφέλιμη θα είναι αυτή η νομοθεσία και στο οικονομικό επίπεδο, στον οικονομικό τομέα. Έχουν διενεργηθεί διάφορες οικονομικές μελέτες που καταδεικνύουν του λόγου το αληθές. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, έχει γίνει υπολογισμός και φαίνεται ότι έξι μονάδες από το ΑΕΠ αφιερώνονται στην κάλυψη δαπανών που έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους θέματα για τους εργαζομένους. Μιλούμε δηλαδή για μια επένδυση η οποία είναι πολύ σημαντική και σε οικονομικό επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνει κανείς παρά να θεραπεύει. Θα πρέπει να δρά πριν προκύψουν τα φαινόμενα για να αποφευχθούν. Η πρόληψη είναι ένα περίπλοκο θέμα το οποίο απαιτεί εποπτεία, κατάρτιση, ε, παρακολούθηση, εκπαίδευση και σχεδιασμό. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε σωστούς κοινωνικούς συνομιλητές, κοινωνικούς εταίρους. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο και δεν θα είχαμε κατορθώσει να εφαρμόσουμε ε, την πρόληψη. Πολύ συχνά λέγεται ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι σίγουρα μικρότερο από το κόστος του θεραπεύειν. Και τέλος, θα ήθελα να, και υπογραμμίσω και τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έρχεται να πει στην κοινή γνώμη, αλλά και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ε, είναι εδώ, είναι παρόν κάτι το οποίο απέδειξε μέσω της πολύ σωστής συνεργασίας τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και ε, του Συμβουλίου και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Σας εύχομαι να συνεχίσετε την ε, συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίνε, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο εν ονόματι της ε, ομάδος, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι σε περίπτωση ψηφίσματος ε, δεν είναι δυνατόν, άρα σήμερα το πρωί μου είπαν ότι πρέπει να παρέμβω τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συζητητές, πράγμα που δεν έκανα προηγουμένως, και τον Στίβεν Χιούς, γιατί ο Στίβεν Χιούς και εγώ το 2004 πήγαμε στα διάφορα νοσοκομεία με τον Τζον Μπόου που ήταν ένας συντηρητικός ε, ευρωβουλευτής και ε, ε, πήγαμε να δούμε δύο διεισόμαση τι συνέβαινε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό διότι εδώ πρέπει να γνωρίζουμε τι χρειάζεται ο επιτόπιος ενδιαφερόμενος και γι' αυτό χρειάστηκε να έχουμε τις απόψεις των ενδιαφερομένων και ο Στίβεν αναφέρθηκε στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και θα ήθελα να γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει ε, εφαρμοστικές ε, κατευθυντήριες γραμμές επί του θέματος που είναι πολύ σημαντικό. Ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου επίσης παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε γιατί είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα προς την εφαρμογή διότι αυτοί οι εργαζόμενοι περίμεναν τόσα χρόνια. Δεν θέλουμε πλέον να υπάρξουν τραυματισμοί περιττή ε, ε, περιμένοντας διότι υπήρξαν υπερβολικά πολύ ε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βεβαίως αυτή τη στιγμή θα μόνο με τον υγειονομικό τομέα αλλά θα ήθελα το ίδιο να γίνει και σε άλλους τομείς και ιδιαίτερα στις φυλακές γιατί είναι βασικό η λειτουργία των φυλακών να μπορούν να προστατεύονται και άλλωστε θα ήθελα να καλύψουμε αυτούς τους εργαζόμενους και επίσης θα πρέπει να έχουμε ε, μία ειδική μνήα στο είδος των βελονών διότι οι διάφοροι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να υπόκεινται υπερβολικούς και άχρηστους ε, τραυματισμούς ε, από, τα, από τέτοιες περιπτώσεις. κυρία Λάμπερτ, σε ευχαριστώ. Σύμφωνο και χαιρετίζω την πράξη αυτή παρόλο που καλό θα ήταν να είχε προηγηθεί διότι έχει ξεκινήσει από το 2001 η κίνηση και επιτέλους μπορούμε να καλύψουμε το θέμα παρόλο που πολλοί έχουν ήδη ε, επηρεαστεί. Ε, όσον αφορά το ε, τους υπολογισμούς θα ήθελα να πω ότι 90% των ε, ε, υπολογισμένων ε, τραυματισμών εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείες ενώ δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση εμφανίζεται ένα ποσοστό γύρω στο 75% σε αυτό το χώρο θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία συμφωνία διότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τα περιστατικά αυτά θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε γιατί δεν ενδιαφέρονται οι, ε, αυτοί οι οποίοι πρέπει να καταρτήσουν τις εκθέσεις και γιατί δεν ενημερώνουν για, αυτές, ε, για αυτούς τους τραυματισμούς ιδίως στους μελλοντικούς τους εργοδότες διότι βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχει και παρακολούθηση όταν υπάρχει μια ενημέρωση δεν υπάρχει παρακολούθηση και ε, δεν υπάρχει ούτε η τεχνική υποστήριξη ούτε η ε, συναισθηματική όταν ε, κάποιος έχει μολυνθεί ή όταν ε, υπάρχει κίνδυνος να μολύνει και άλλους ασθενείς αν έχει μολυνθεί με τον ιό του AIDS. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με τις αντιδράσεις των εργοδοτών. Πολλοί έχουν αναφερθεί στο θέμα αυτό και γι' αυτό πρέπει να καλύψουμε και τους μαθητευόμενους, τους υπεργολάβους, το προσωπικό καθαρισμού. Γι' αυτό δεν είμαι πολύ βέβαιη, αλλά θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να καλύπτουμε ε, και τους εργαζόμενους στους άλλους τομείς οι οποίοι εμπλέκονται. Είναι πολύ βασικό θέμα. Ελπίζω ότι ε, θα πρέπει ε, τα κράτη να αντιληφθούν ότι χρειάζεται υποχρεωτική επιμόρφωση, ιδίως ε, ε, για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιμόρφωση ακόμη και όταν οι εργοδότες έχουν εγκαταστήσει τέτοιες πολιτικές. Επίσης ε, η πρόληψη και η επιμόρφωση θα καλύψουν το 1 τρίτον από το κόστος που καταβάλλεται τώρα για την θεραπεία από τραυματισμούς με αιχμηρά αντικείμενα πράγμα το οποίο θα είναι ισόφελος ε, και των εργοδοτών οι οποίοι ε, θα κινδυνεύουν με ε, προσφυγές νομικές εάν δεν έχουν λάβει μέτρα. Ο κύριος Βλάζακ τώρα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η συμφωνία πλαίσιο για την πρόληψη των τραυματισμών στο νοσοκομιακό τομέα. Είναι η πρώτη συμφωνία που έχει συναφθεί από Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Οργάνωση και είναι σημαντικό που συνέβη αυτό γιατί έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο περιστατικά το χρόνο. Αν γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία θα Σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας και θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στο νοσοκομιακό περιβάλλον από τέτοιου είδους τραυματισμούς. Υπάρχουν ναι μεν κάποιες ασάφειες στους ορισμούς της ίδιας της συμφωνίας, πιστεύω όμως ότι θα καταβληθούν όλες οι προσπάθειες έτσι ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να μας παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τελικά και το Συμβούλιο να μπορέσει να υιοθετήσει αυτήν την οδηγία. Τονίζω ότι μια συμφωνία ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό μέσο που είναι άνευ προηγουμένου σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η μορφή αυτορύθμισης που συνάπτεται μέσω συμφωνίας από τους άμεσα ενδιαφερομένους είναι εξαιρετικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής αυτορύθμισης. Δεν είναι εντελώς αντίθετο από ε, την, ε, το σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα όπου πολλές εταιρείες πρέπει να ανεχθούν την νομοθεσία που τους επιβάλλουμε εμείς. Κύριος Μαστάλκα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να, να ευχαριστήσω τους τις εισηγήτριες για τις εξαίρετες προσπάθειές τους για την, το κείμενο αυτό. Εγώ ο ίδιος είμαι ιατρός και χαίρομαι ιδιαίτερος που εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο συνειδητοποιούμε την ανάγκη για μια καλύτερη προστασία των εργαζομένων στο νοσοκομιακό τομέα από τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα. Αυτό πάντως που με ανησυχεί είναι ότι υπάρχει καθυστερημένη πρόοδος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που επιστήσαμε το, την προσοχή της Κομισιόν στο θέμα αυτό και ακόμα περισσότερα από το ψήφισμα της, ε, του Κοινοβουλίου όπου ζητούμε νομοθετικό κείμενο για την προστασία των εργαζομένων στο νοσοκομιακό τομέα. Στο προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου συνεργάστηκα με την κυρία Λίν και και αυτό λοιπόν Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω το ταχύτερο δυνατό να υιοθετηθεί το σχέδιο οδηγίας και θα ήθελα να έχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία για τους εργαζομένους. Κυρία Μωράν Σαχτιέ, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερος διότι σήμερα το πρωί έχουμε επιτέλους αυτή την πρόταση οδηγίας για την πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα. Και χαίρομαι ιδιαίτερο, διότι πρόκειται για ένα πρόβλημα υγείας το οποίο οφείλουμε να λύσουμε το συντομότερο δυνατό, διότι γνωρίζουμε όλοι πόσο δραματικές είναι οι συνέπειες από αυτούς τους τραυματισμούς. Και θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να σας πω ότι εμπιστεύομαι πλήρως ε, την ε, εσάς και τον τρόπο με τον οποίο θα δράσετε, γιατί η λύση που προτείνετε θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια κύρια Λίν και τον κύριο Γιούξ, γιατί πράγματι δική μας ευθύνη ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να κάνουμε το παν για την προστασία των συμπολιτών μας. Βεβαίως εδώ ε, το θέμα αφορά τους επαγγελματίες της υγείας, αφορά όμως και το προσωπικό που εργάζεται στην καθαριότητα, τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά και το προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία, στην εκπαίδευση. Ουσιαστικά αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν θα πρέπει να κάνουν αυτούς που τους φροντίζουν να διακινδυνεύουν ε, την υγεία τους. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι βεβαίως και θα κινητοποιηθούμε, θα υποστηρίξουμε τους εισηγητές για να εφαρμοστεί στο σύνολό του το νομικό αυτό μέσο σε όλα τα κράτη-μέλη και σίγουρα θα οργανώσουμε συνεδριάσεις όπου θα έχουμε ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά. Είναι δική μας δέσμευση, είναι δική μας ευθύνη, ε, αφορά όλους και θα πρέπει όλοι να ασχοληθούν. Ευχαριστώ κυρία Ράπτη, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους παλαιότερους συναδέλφους που βρήκα στο Κοινοβούλιο, που βρίσκομαι για πρώτη θητεία, τον καλό συνάδελφο κύριο Χιούς, την κυρία Λίν, την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές, γιατί βρήκα μια έτοιμη δουλειά για ένα θέμα το οποίο με κάποιο τρόπο με αφορά και προσωπικά. Ο άντρας μου είναι γιατρός και πριν από μερικά χρόνια μολύνθηκε από μια βελόνα άρα ξέρω πολύ καλά την αγωνία που αισθάνεται μια οικογένεια ενός εργαζόμενου σε νοσοκομείο που τραυματίζεται από αιχμηρό αντικείμενο. ήταν πραγματικά δύσκολες οι μέρες που πέρασαν περιμένοντας να δούμε τα αποτελέσματα έτσι λοιπόν θέλω πραγματικά για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχει γίνει αλλά να εκφράσω και την ικανοποίησή μου που για πρώτη φορά βλέπουμε οργάνωση εργοδοτών και οργάνωση εργαζομένων να συμπράττουν να συμφωνούν και να καταλήγουμε σε αυτό το ψήφισμα. αισθάνομαι ότι πραγματικά η ευρωπαϊκή ένωση πραγματώνει τους στόχους της λαμβάνοντας πια αποφάσεις με τους πολίτες της για τους πολίτες της θυμίζω κάτι που επανέλαβαν και άλλοι συνάδελφοι αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία του να το λέμε και να το θυμόμαστε συνεχώς ότι ένα εκατομμύριο ε, τραυματισμοί από αιχμηρά αντικείμενα συμβαίνουν. δεν μπορώ να μην, υπερτονίσω το ρόλο που έχει παίξει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το οποίο από το 2005 εργάζεται σοβαρά για αυτήν την υπόθεση με δεδομένη από την άλλη πλευρά την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει μια έλλειψη που είναι ιδιαίτερα έντονη και στην πατρίδα μου την ελλάδα σημειώνω ότι θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πολύ γρήγορη εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος αυτής της οδηγίας. πρόκειται για μια απόφαση που θα συμβάλλει εκ των πραγμάτων και στους κοινωνικούς στόχους της ευρωπαϊκής ένωσης που ανάμεσά τους βρίσκεται η αύξηση της απασχόλησης θυμίζω πως η ευρωπαϊκή επιτροπή δήλωσε πρόσφατα σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο διαστόματος του επανεκλεγέντος προέδρου της πως ένας από τους τομείς στους οποίους στοχεύει να επενδύσει είναι και οι λεγόμενες λευκές θέσεις εργασίας. ας σώσουμε λοιπόν ζωές και κυριολεκτικά και μεταφορικά δημιουργώντας σε αυτήν την τόσο δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά περίοδο πολύτιμες θέσεις εργασίας. τελειώνοντας θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη δουλειά του νέου επιτρόπου και αν μου επιτρέπετε να πω το εξής ο εκλεκτός και έμπειρος συνάδελφος κύριος Σέρκας σας είπε προηγουμένως ότι εύχεται να μπείτε και να συνεχίσετε με το δεξί. εγώ εύχομαι να μπείτε και να συνεχίσετε με το αριστερό και το λέω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσέγγιση που θα φέρει το κοινωνικό πρόσωπο της ευρώπης στην επιφάνεια. το νου σας το μυαλό σας στους εργαζόμενους. το έχει ανάγκη ο ευρωπαϊκός λαός. ευχαριστώ. Και εγώ θα σας παρουσιάσω την προσωπική μου εμπειρία. Δεκαπέντε χρόνια εργαζόμουν στο νοσοκομείο και μάλιστα και ως παρασκευάστρια σε χειρουργείο. Και μένα έχει συμβεί να έχω τραυματιστεί από αιχμηρά αντικείμενα. Και όπως είπε και η κυρία Ράπτη, ε, ακόμα θυμάμαι το άγχος μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Και υπάρχει ένα παράθυρο ανάμεσα στην μόλυνση και στην ε, εκδήλωση της ασθένειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το υιοθέτηση της ε, του κειμένου για να έχουμε ελάχιστα πρότυπα για όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομιακό τομέα. Είναι το 10% του εργατικού δυναμικού το νοσοκομιακό δυναμικό στην Ευρώπη και έχουμε δύο εκατομμύρια τραυματισμούς και συχνά συχνά υπάρχει ε, αποθάρρυνση του προσωπικού και εγκατάλειψη αυτού του εργασιακού περιβάλλοντος. Το 2,5% των περιπτώσεων θα μπορούσαν να γίνουν AIDS ή 40% των περιπτώσεων να οδηγήσουν σε υπατήτηδα Β ή Γ. Ο... Μάλιστα το ίδιο το επάγγελμα εξαιτία αυτών δεν είναι ελκυστικό. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος για τις μεμονωμένες νοσοκομιακές μονάδες και εξετάζοντας Όλα αυτά τα πρωτόκολλα που χρειάζονται έξι μήνους για να εφαρμοστούν είναι προφανές ότι αυξάνεται το κόστος για όσους έχουν μολυνθεί από ασθένεια. Εφόσον λοιπόν ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί, είναι απαραίτητο να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν τα μέτρα και οι εργαζόμενοι να τα σεβαστούν. Thank you. Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε ένα πρόβλημα το οποίο όντως αυξάνεται και θα γίνει ένα από τα πολύ βασικά θέματα εις ε, το χώρο. Ε, αλλά αναφέρομαι εδώ στις στατιστικές, διότι εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μιλάμε για ένα εκατομμύριο και σε παρεμφερείς καταστάσεις ε, ε, σε παρεμφερείς καταστάσεις τέτοιων ατυχών τραυματισμών ενώ στην Αμερική έχουμε 380.000 ε, παρεμφερεί περιστατικά. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ε, εργαζόμενοι αλλά υπάρχουν και οι ασθενείς οι οποίοι υφίστανται την, τον ίδιο κίνδυνο και αυτό οδηγεί σε πολύ μεγάλες αποζημιώσεις οι οποίες πρέπει να καταβληθούν από τα νοσοκομεία προηγούμενοι ομιλητές είπαν ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το τομέα διότι η πρόληψη είναι αυτή η οποία είναι φθηνότερη από την ε, θεραπεία. Το ψήφισμα αυτό όντως αξίζει να υποστηριχτεί και ε, είναι ένα από τα θέματα τα οποία ε, μας έχουν ζητηθεί από τον υγειονομικό τομέα αλλά και οι αποζημιώσεις που πληρώνουν τα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί ε, η υγειονομική ε, λειτουργή τις απαιτούν και αυτό το ποσό είναι σημαντικό η πολιτική μου ομάδα στηρίζει αυτή, αυτό το ψήφισμα διότι πιστεύω ότι μέσω αυτού θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ορισμένες προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα και να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών και, των, και του προσωπικού. Κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω σήμερα το λόγο για να ε, συγχαρώ καταρχάς όλους τους εισηγητές και όλους όσους ε, προκάλεσαν αυτή τη συζήτηση. λέμε κάποιες φορές ότι η ευρώπη πρέπει να έρθει πιο κοντά στους πολίτες. με αυτή τη συζήτηση πραγματικά το καταφέρνουμε. συζητούσα με φίλο μου συνομήλικο δικό μου νέο ειδικευόμενο γιατρό και όταν του μετέφερα αυτή τη συζήτηση εκείνος με ιδιαίτερη χαρά μου είπε ότι πράγματι αυτό είναι καθοριστικό και προσπαθήστε να εξηγήσετε σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες τι ακριβώς κάνετε. είναι σημαντική η πρόληψη ε, και η ενημέρωση όλων όσων εργάζονται στα νοσοκομεία σε σχέση με τους κινδύνους που διατρέχουν και είναι πράγματι καθοριστικό να ε, εξηγήσουμε σε όλους ότι όταν εργάζονται με τόσο πιεσμένα ωράρια ότι όταν οι χώροι καμιά φορά είναι μικροί όταν οι ασθενείς είναι πάρα πολλοί είναι καθοριστικό να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί τουλάχιστον να μπορούν να λαμβάνουν τα περισσότερα και απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χρειαζόμαστε υγιές προσωπικό που εργάζεται στα νοσοκομεία προκειμένου και εμείς ως ασθενείς κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή, την καλύτερη δυνατή ε, το, καλύτερο, το, ενδιαφέρον τους και την καλύτερη δυνατή φροντίδα από εκείνους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. And now, Mrs. Kadenbach for one minute. Ευχαριστώ. Κυρία Κάντενμπεργκ για ένα λεπτό. Στην πολιτική μας πρέπει να είναι στόχος να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους και ε, για, σε αυτό συμβάλλει και η δημιουργία θέσεων εργασίας χωρίς να ξεχνάμε ότι οι θέσεις αυτές εργασίας δεν πρέπει να καθιστούν άρρωστους τους ανθρώπους ή να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους γι' αυτό και θα πρέπει να θεωρήσουμε πολύ βασικό και την, ε, τις θέσεις εργασίας αλλά και τη διατήρηση της υγείας. Πιστεύω ότι αυτή η ρύθμιση ε, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό διότι ε, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό καθημερινά. Γι' αυτό και κάθε Ευρωπαίος και κάθε Ευρωπαία προφανώς απαιτεί να εφαρμοστεί για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους σήμερα και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι για την ευρεία υποστήριξη για την πρόταση αυτή στο Κοινοβούλιο. Λυπάμαι γιατί η όλη διαδικασία διήρκησε πολύ περισσότερο από όσο περιμένατε, αλλά είμαι πεπισμένος ότι ο κοινωνικός διάλογος έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση των κοινωνικών εταίρων. Δεν βοηθάει μόνο την νομιμότητα της απόφασης, αλλά και την εφαρμογή της, γιατί όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία των νέων κανόνων ενδιαφέρονται και στην επιτυχία τους. Και αυτό είναι σημαντικό. Ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για κάποιες διευκρινήσεις για την αποσαφήνιση της συμφωνίας πλαίσιος και για την εφαρμογή της. Ελπίζουμε λοιπόν και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την τελική θέση και του Συμβουλίου και αυτό θα απαντήσει και σε κάποιες από τις ανησυχίες για την εφαρμογή για την μακροχρόνια παρακολούθηση τώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε το πόσο επιτυχής θα είναι αυτή η νέα οδηγία. Εφιστώ την προσοχή σας στο κείμενο που λέει ότι συμβαλόμενα μέρη θα αναθεωρήσουν την εφαρμογή αυτής της ομφυνίας πέντε χρόνια μετά από την ημερομηνία της έσωσης εάν το ζητήσει η μία από τις δύο συμβαλόμενες πλευρές. Είναι δηλαδή σημαντικό αυτό. Υπάρχει παρακολούθηση της συμφωνίας και εάν υπάρχει αλλαγή στον αριθμό των περιστατικών των τραυματισμών. Τέλος, είναι η δεύτερη μου μέρα ως νέος επίτροπος και Κάποιοι ομιλητές το τόνισαν αυτό στις παρεμβάσεις τους. Πράγματι, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στους ξεχασμένους της Ευρώπης, σε αυτές τις ηλικιακέ ομάδες, σε αυτούς τους ευάλωτους που δεν μπορούν εύκολα να μιλήσουν μόνοι τους και οι οποίοι συχνά αγνοήθηκαν και παραμερίστηκαν σε προηγούμενες εποχές. Ο νοσοκομιακός τομέας σαφώς και είναι πολύ σημαντικός τομέας. Πρέπει να υπάρχει αφοσίωση και προσοχή. Και δεν είναι μόνο ότι είναι εκτεθειμένοι σε αιχμηρά αντικείμενα και μολύνσεις. Ξέρουμε ότι εργάζονται πολύ μεγάλες και μακριές ώρες. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πολύ ολοκληρωτική προσέγγιση να προσέξουμε τέτοιου είδους ομάδες που είναι πολύ σημαντικές ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεων όταν η αναμενόμενη δημοσιονομική μείωση θα επηρεάσει αυτές τις ομάδες. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της προσοχής, της μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση. Και ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.